Allora Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής μας. Χθες το απόγευμα, με ακούτε, διακόπτει ο πρόεδρος. Χθες το απόγευμα λοιπόν η Επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ψηφοφορία στο καθεστώς χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, αφήνοντας όμως ανοιχτή την δυνατότητα να συνεχιστεί η συζήτηση επί της ουσίας. Νομίζω ότι θα έρθει η κυρία Γιαννάκου όπου να είναι. Η ψηφοφορία θα αναβληθεί για μια έκτακτη συνεδρίαση μας, η οποία θα μπορούσε να είναι πριν από την επόμενη ολομέλεια του Στρασβούργου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Μόλις τώρα φτάνει η κυρία Γιαννάκου. Λοιπόν, οι ψηφοφορίες μας θα είναι πάρα πολύ απλές συνεπώς. Αφορούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διατάξεως, την επιστολή δηλαδή, για την ερμηνεία του άρθρου 159 του κανονισμού. Ήδη χθε συζητήσαμε το τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοψηφίας στις περιπτώσεις πρότασης προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπήρξε ε, συμφωνία για να υπάρξει μια επιστολή. Θέτω σε ψηφοφορία την επιστολή. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά της επιστολής. Λοιπόν, ποιοι είναι κατά παρακαλώ. Αποχές. Καλώς γίνεται δεκτή η πρόταση επιστολής με τη δική μας ερμηνεία του άρθρου 159. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τώρα αυτά που συζητήσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συντονιστών. Πήραμε τις εξής αποφάσεις σχετικά με τις εκθέσεις που θα σας προτείνουμε βέβαια προς έγκριση. Εκθέσεις πρωτοβουλίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε άνω των έξι σε εξέλιξη μέχρι πέντε κανονικά, αποφασίσαμε να ζητήσουμε να υπάρξει δυνατότητα και για μία έκτη σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις για τις εκλογές του 2014. Η συγητής μας είναι ο κύριος Νταφ. Υπήρξαν άλλες δύο προτάσεις δεν μπορούμε να τις καταθέσουμε επίσημα. Τη μία θα προσπαθήσουμε να την προωθήσουμε όταν ολοκληρωθεί <clears throat> συγγνώμη, η πορεία μίας ε, ε, από τις πέντε πρώτες εκθέσεις. Όταν κλείσει μία από τις πέντε θα μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα της εφαρμογής σε επίπεδο θεσμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο επί τη βάση του άρθρου 11 από ό,τι φαίνεται θα ζητήσει να υπάρξει μια διαδικασία διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο για την τροποποίηση της εκλογικής πράξης έτσι ώστε οι εκλογές ε, το 14 να γίνουν τον μήνα Μάιο, ένα μήνα νωρίτερα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα για την ε, πρόταση αυτή και να γνωμοδοτήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. ταυτόχρονα δώσαμε στη σοσιαλιστική ομάδα την πρόταση τροποποίησης του 116.2 του κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων της 17ης Ιανουαρίου του 2013. Επιβεβαιώσαμε επίσης την επίσκεψη στο Λονδίνο μιας αντιπροσωπείας μας στις 19 και 20 Ιουνίου. Επιβεβαιώσαμε παράλληλα ότι μια αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην πόλη της Ουάσιγκτον τον επόμενο Οκτώβριο. 27, 28, όχι, 28 με 31 Οκτωβρίου ο πρόεδρος, δύο μέλη του ΕΛΚ, δύο μέλη των σοσιαλιστών και από ένας από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Ζητήσαμε επίσης να ζητήσουμε την αδειοδότηση μιας μήνυα ακροάσεως για τις έδρες Ευρωπαϊκό, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγητές εδώ είναι δύο, ο κύριος Φόξ και ο κύριος Χέφνερ θα πρέπει να κάνουν τις προτάσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο ε, της ε, ακροάσεως και τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων. Περιμένουν φυσικά ε, προσφορές εισαγωγικά και από πλευράς των σκιωδών εισηγητών και κυρίως των συντονιστών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί σε επίπεδο συντονιστών. Δεν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από ό,τι καταλαβαίνω από πλευρά σας. Καλώς. Λοιπόν, στην παρούσα φάση, μιας και είναι ανάμεσά μας πλέον η κυρία Γιαννάκου, θα ήθελα να περάσουμε στην συζήτηση εκ νέου το θέματος ε, του καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η κυρία Γιαννάκου είναι γνώση ότι χθε η Επιτροπή μας αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ψηφοφορία της εκθέσεώς της, αλλά να εμείνουμε λίγο περισσότερο στο περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής. Ευχαριστώ την κυρία Γιαννάκου για την παρουσία της εδώ ε, να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να μείνουμε στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε αποφασίσει για τις ψηφοφορίες. Γνωρίζω ότι η κυρία Γιαννάκου χρειάστηκε να κάνει πολλές αλλαγές στο πρόγραμμά της για να είναι παρούσα, αλλά αντί για την ψηφοφορία θα μπορέσουμε να έχουμε μια χρήσιμη συζήτηση, λοιπόν. πάνω σε αυτό το σχέδιο εκθέσεως ε, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Δεν ξέρω, μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου, να κάνετε μια εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εφόσον ε, ε, οι πολιτικές ομάδες έχουν διαφοροποιηθεί και έχουν αλλάξει στάση και θέλουν να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι η χθεσινή απόφαση δεν είναι νόμιμη. Με 7 μέλη παρόντα δεν είναι νόμιμη η απόφαση. Οφείλω να το επισημάνω αυτό. Διότι κύριε Πρόεδρε χρειάζεται και κάποια δεοντολογία στην Επιτροπή. Δεν μπορούν οι πολιτικές ομάδες να αλλάζουν όποτε τους αρέσει θέση. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Την προηγούμενη φορά στη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο ανέφερα, διότι αυτό είναι μόνο το θέμα το ανοιχτό. Δεν είναι όλα τα θέματα ανοιχτά. Το μόνο ανοιχτό θέμα είναι ότι περιμέναμε την legal opinion της Επιτροπής ε, του νομικού τμήματος του Κοινοβουλίου για να τοποθετηθούμε επ' αυτού και να δούμε πώς θα φτιάξουμε την... Ε, ε, τροπολογία συμβιβασμού. Εγώ σας ανέφερα στο Στρασβούργο ποια είναι η δική μου θέση σε σχέση με αυτά που λέει ε, η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και νομίζω και είμαι ε, πραγματικά στη διάθεσή σας να ακούσω πώς τοποθετούνται τα μέλη έναντι αυτού του θέματος. Διότι επαναλαμβάνω, δεν θα αρχίσουμε τη συζήτηση από την αρχή, την έχουμε εξαντλήσει. Το θέμα που είχαμε να συζητήσουμε είναι αυτό για το οποίο απευθύναμε ερώτημα στη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, πώς διαρθρώνονται τα κόμματα και ποιοι μπορούν να, κάνουν, να δημιουργήσουν κόμμα, πώς κρίνεται το θέμα εάν υπάρχουν παράπονα εναντίον ενός κόμματος και ποιος το κρίνει και όλο αυτό το τμήμα το οποίο ήταν και το επίμαχο. Δηλαδή υπήρχαν ερωτηματικά επ' αυτού. Εγώ λοιπόν είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις απόψεις όλων. Έχω εκφράσει τις απόψεις μου και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τις επαναλάβω. Ήμουνα πολύ συγκεκριμένη στο Στρασβούργο στη συνάντηση που είχαμε. Κύριε κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει να κάνουμε είναι καταρχάς να πούμε ότι στο Στρασβούργο χάσαμε τον περισσότερο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, υπήρξε μια κάποια σύγχυση. Είναι σαφές ότι θα ψηφίσουμε στο επόμενο Στρασβούργο, είναι σαφές ότι μπορούμε να τελειοποιήσουμε, αν θέλετε, τις συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες έχει κάνει η φίλη Μαριέτα και η Σκιώδης και θα πρέπει πολύ σύντομα να ασχοληθούμε με το θέμα της άποψης της νομικής υπηρεσίας. Έχουμε λοιπόν τις συμβιβαστικές, έχουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις ε, νομικές απόψεις κάποιων άλλων οργάνων και αν υπάρχουν διαφορές ε, θα πρέπει να επιλέξουμε. Κατανοώ αυτό που είπε η κυρία Γιαννάκου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρξει μια νέα γενική συζήτηση που έχουν γίνει οι συζητήσεις αυτές. Μόνο κάποιες αλλαγές για τις συμβιβαστικές, ε, πιθανώς τις συμβιβαστικές και πέραν αυτού ουδέν. Πρέπει να κλείσει η συζήτηση. Έχουν συζητηθεί συμβιβαστικές προτάσεις μέχρι τώρα αρκετά αναλυτικά και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ψηφοφορία Έχουμε εξαντλήσει τις συζητήσεις που έπρεπε να κάνουμε και απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να μην ανοίξουν εκ νέου τις συζητήσεις πάνω στις συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουμε ήδη καταλήξει. Ξέρω ότι κάποιοι από σας ε, το ζήτησαν αυτό στο Στρασβούργο, αλλά η συζήτηση περιορίστηκε ουσιαστικά στο θέμα του χρονοδιαγράμματος τότε. Ας ε, κλείσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα και ας προετοιμαστούμε σωστά για την ψηφοφορία που δεν θα πρέπει να αργήσει. Κύριος Νταφ. Κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι είναι σωστό αυτό που είπαμε, να αναβάλουμε την ψηφοφορία δηλαδή. σε, σεβόμεθα τις προσπάθειες που έχουν γίνει, αλλά υπάρχει ακόμα ένα κάποιο περιθώριο προπαρασκευής των πολιτικών ομάδων, εφόσον θέλουμε να είμαστε συνεκτικοί. Πήραμε τα τελικά στοιχεία χθε το απόγευμα και πολλές από τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες θα πρέπει σαν παράδειγμα να διαιρεθούν Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια κάποια προσπάθεια και αν συνεχίζαμε απευθεία στην ψηφοφορία σήμερα, αυτό θα προκαλούσε μια κάποια σύγχυση και μια κάποια έλλειψη οργάνωσης, θα έλεγα. Δεύτερον, έχουμε τρεις νομικές νομοδοτήσεις. Καμία δεν συμφωνεί με την άλλη. Αυτό και μόνο νομίζω απαιτεί, επιβάλλει την περαιτέρω εξέτασή τους. Τρίτον, στα θέματα ουσίας και αναφέρθηκα σε αυτά στο Στρασβούργο, υπάρχουν τρία θέματα, τρία θέματα τα οποία απαιτούν περισσότερη συζήτηση. Πρώτον, το θέμα της νομικής προσωπικότητας στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Τι θα συνεισφέρει στην αυτονόμηση των πολιτικών αυτών ε, κομμάτων στα πλαίσια της προσπάθειας ε, ε, των προεκλογικών εκστρατιών και ανταγωνιζόμενα τα κόμματα αυτά πολλές φορές τα εθνικά τους κόμματα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ουσία. Παρά το ότι εμείς αναγνωρίζουμε την αυτόνομη νομική προσωπικότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος, παρόλα αυτά τα κόμματα αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε κάποιον εθνικό νόμο ή σε κάποια σύνθεση εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια δημιουργίας ενός αυτονόμου νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, κάτι το οποίο δεν έχουμε ολοκληρώσει. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ο πλήρης διαχωρισμός της δυνατότητας καταγραφής του πολιτικού κόμματος. Είναι μια τεχνική διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην τεχνική καταγραφή και την πολιτική αξιολόγηση η οποία μπορεί να έχει σχέση με την παραβίαση βασικών αξιών κτλ. Συμφωνούμε νομίζω αρκετοί εδώ λέγοντας ότι η διατύπωση στο αρχικό κείμενο γύρω από τα θέματα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη, δεν είναι ιδιαίτερα επακριβής μάλλον. Και τρίτο θέμα αφορά στην οργάνωση του ιδίου του Κοινοβουλίου. Τι ακριβώς όργανο είναι το Κοινοβούλιο, ε, ποιο είναι το όργανο του Κοινοβουλίου, το οποίο θα είναι ε, υπεύθυνο για την καταγραφή πρώτον των κομμάτων και δεύτερον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίζουν εάν έχει υπάρξει μια παραβίαση των αξιών και των αρχών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε ένα τομέα στον οποίο θα πρέπει να είμαστε ε, πιο συγκεκριμένοι σε επίπεδο διακανονισμού. και σε σχέση με τις κυρώσεις, τις ποινές, τα πρόστιμα κτλ. που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες στην περιγραφή τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, ε, ε, καλείται να εφαρμόσει τον κανονισμό ή να ζητήσει την εφαρμογή ενός κανονισμού, αλλά δεν είναι σε θέση να ελέγξει απόλυτα ή να επιβάλλει την εφαρμογή ενός κανονισμού. Πρέπει λοιπόν εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, θα έλεγα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι με λίγες συντομότατες συζητήσεις πάνω στα τρία θέματα που προανέφερα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε βελτιωμένες συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια διακομματική συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Ντάφο, κύριος Μπρόνς. Uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν ζητώ συγγνώμη που συμπεριφέρθηκα καταλήλως ε, χτες ε, γιατί ήρθα και δεν ανάγκασα αρκετούς ε, να έρθουν ώστε να έχουμε απαρτία. Ε, πραγματικά ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά. Δεύτερον, μας είπαν ότι δεν θα πρέπει να μιλήσουμε για τις τροπολογίες που ήδη έχουν συζητηθεί. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για την τροπολογία που δεν έχει κατατεθεί, αλλά υπονοείται σε ολόκληρη την έκθεση. Στην ε, τροπολογία Α και στην αρχική διατύπωση λέει, ορίζει ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Και η αρχική διατύπωση αλλά και η συμβιβαστική Α το ορίζουν ως ε, μία πολιτική συμμαχία που επιδιώκει πολιτικούς στόχους. Εγώ πιστεύω πως η τροπολογία που έπρεπε να έχει κατατεθεί είναι η προσθήκη των λέξεων εγκεκριμένη από την πολιτική τάξη που, ε, θα ακολουθεί δηλαδή τη λέξη στόχους. Ένα πολιτικό, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα είναι ε, μια πολιτική συμμαχία που επιδιώκει πολιτικούς στόχους που εγκρίνονται από την πολιτική τάξη. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν την τροπολογία που δεν έχει κατατεθεί. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητά το λόγο. Κύριε Σκούζα. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω για τη διαδικασία ότι θεωρώ σωστό να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που μας είναι απαραίτητος. Και εχθές Συζητήθηκε το θέμα, πήραμε μια απόφαση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις συμβιβαστικέ προτάσεις, ποιες μπορεί να δεχτεί η συγγήτρια, ποιες όχι και κατόπιν να συμφωνήσουμε στις πολιτικές ομάδες. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή έκθεση που αφορά τις μελλοντικές ε, πολιτικές προοπτικές και έχει σημασία για την Ευρώπη του μέλλοντος. Θα ήθελα επίσης να πω στον συνάδελφο ότι είμαστε βεβαίως ε, όλοι πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να δούμε τη διατύπωση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή λέμε ότι τελικά θέλουμε η αναγνώριση του τι είναι ή του τι δεν είναι κόμμα ή ότι κάποια πολιτική ε, δύναμη είναι κόμμα, θα πρέπει να λαμβάνεται σε τελική ε, βαθμίδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό νομίζω ότι είναι η άποψη της πλειοψηφίας αυτής της Επιτροπής και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια τέτοια συμβιβαστική πρόταση, αλλά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη η διατύπωση εδώ, να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση. τελικά μετά την αν θέλετε απόφαση σε περίπτωση αμφιβολίας υπάρχει το Κοινοβούλιο, υπάρχει το Συμβούλιο, υπάρχει η Επιτροπή, είμαστε οι τρεις οι εκπρόσωποι των τριών θεσμικών οργάνων που μπορούμε να ε, αποφασίσουμε. Αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η τελική, αν θέλετε, βαθμίδα και ουσιαστικά θα πρέπει να πρόκειται για ανεξάρτητους, αν θα πρόκειται για μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, αν θα πρόκειται για εμπειρογνώμονες εξωτερικούς, οι οποίοι όμως θα διορίζονται από τα τρία θεσμικά όργανα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξαναεπεξεργαστούμε αυτό το σημείο, γιατί είναι καθοριστικό, είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό, μια σημαντική, αν θέλετε, ε, απόφαση και θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση. Δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα επίσης να αναφέρω, έχουμε τις προτάσεις της εισηγήτριας όσον αφορά τις ε, τροπολογίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την βάση χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε την πρόταση το 85%, 15%. Ξέρω ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν εκφραστεί, αλλά τελικά ξέρω ότι συμβιβασμός δεν βρέθηκε για αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις απόψεις, φαίνεται να υπάρχει ακόμα διαφορά μεταξύ της πρότασης της και των διαφόρων προτάσεων των πολιτικών δυνάμεων. Εδώ υπάρχει δυνατότητα να βρούμε έναν συμβιβασμό. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην συμβαστική τροπολογία H. στην τωρινή διατύπωση, στην πιο πρόσφατη διατύπωση αυτής της, συμφων... αυτής της συμβαστικής τροπολογίας, διαβάζω «Promotion of balance of gender». Δεν βρίσκω το κείμενο, αλλά νομίζω ότι εδώ η διατύπωση, έχω σημειώσει, θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί. Να μιλήσουμε δηλαδή για ίσες ευκαιρίες. Να μιλήσουμε για δικαιοσύνη, ίση εκπροσώπηση. Σκοπός μας είναι εδώ να διασφαλίσουμε την σωστή εκπροσώπηση των γυναικών. Να εκπροσωπούνται εξίσου και οι γυναίκες. Ίσως λοιπόν εδώ κάτι μπορούμε να κάνουμε. Να τους δώσουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία. Γιατί αν δεν κάνουμε κάτι εδώ, ακόμα κι αν υπάρχουν οκτώ γυναίκες υποψήφοι σε μία λίστα, αν οι τέσσερις πρώτοι, αυτοί δηλαδή που εκλέγονται είναι άνδρες, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να ξαναδούμε εδώ το αν υπάρχουν γυναίκες σε εκλέξιμες θέσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε λοιπόν και τη διατύπωση αλλά και αυτά τα θέματα τα οποία τα θεωρώ ουσίας. Eh, Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο συνάδελφος Γκέραϊρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να κάνω μια γενική διαπίστωση. Θα πρέπει στην επόμενη συνεδρίασή μας να ψηφίσουμε. Θα έχουν γίνει αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, τα επίπεδα συζήτησης, περάσαμε από διάφορα στάδια, προσπαθήσαμε να τελειοποιήσουμε και θα τελειοποιήσουμε ακόμα την τελική πρόταση για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου του μηνός Απριλίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε παρακαλώ να αναφερθώ στην συμβιβαστική παρίθμου 2 παρακαλώ. Ε, συγγνώμη, ε, δέλτα. Στο τρίτο σημείο αυτής της συμβιβαστικής λοιπόν υπάρχει μία αναφορά στις βασικές αξίες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ισότητα κτλ. Είναι αλήθεια ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η πρόταση, αυτή η διαπίστωση έχει ήδη ενταχθεί στο σημείο ένα της ίδιας τροπολογίας, η οποία αναφέρεται στο δεύτερο άρθρο, στο άρθρο υπαριθμών 2 της συνθήκης. Εγώ νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι καλό να διατηρήσουμε το C αγγλικό, αναφερόμενοι πάντα στο άρθρο 2. Έχει γίνει ήδη μια συζήτηση επί της ουσίας στην Επιτροπή μας. Αν κάνουμε μια αναφορά στη συνθήκη της Ένωσης, στηρίζουμε τις αξίες ακριβώς στην διατύπωση <clears throat> τη συνθήκης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αυτή την δυνατότητα σε όσους έχουν αντιρρήσεις στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφύγουν σε αυτά τα οποία επιβάλλει η συνθήκη. Ενώ αν διατηρήσουμε το σημείο C, νομίζω ότι αναφερόμαστε σε καθολικές αξίες, σε παγκόσμιες αξίες, οι οποίες Υπάρχουν μεν στη συνθήκη, αλλά προϋπήρχαν τις συνθήκες. Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις αξίες οι οποίες προϋπήρχαν και ήταν καθιερωμένες και σεβαστές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι αναζητούν μια θα έλεγα δυνατότητα καθιέρωσης του πολιτικού προτύπου του ευρωπαϊκού να στηριχθούμε όχι σε μία απλή αναφορά, σε μία συνταγματική ρύθμιση όπως είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά σε μία ευρύτερη καθολική αξία. Ευχαριστώ, συνάδελφος Τσακώσκη. Εγώ νομίζω πως όσον αφορά την ψηφοφορία συμφωνούμε ότι θα ψηφίσουμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Δεν γίνεται συντομότερα. Ο, τώρα όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες και το γενικότερο πνεύμα, γιατί πολλοί το συζητούν αυτό, ε, θα ξεκινήσω από την αρχή. Νομίζω πως το πρόβλημα με την καταγραφή των, των ε, πολιτικών κομμάτων ότι δεν θέλαμε να γίνει εξαιρετικά πολιτική φύση αυτή η διαδικασία. Η Κομισιόν θέλει να το κάνει ειδική το Ευρωκοινοβούλιο και καταλαβαίνουμε γιατί η αρχική μα αντίδραση ήταν ε, τουλάχιστον να μοιράσουμε την ευθύνη με το δικαστήριο γιατί όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό με αμερόληπτο τρόπο. Στην αρχή ορισμένοι δεν ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με το θέμα της Επιτροπής Σοφών, ακούσαμε όλα τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω πως έχουμε ξεπεράσει εκείνο το σημείο, δηλαδή ότι η Επιτροπή Σοφών θα πρέπει να υπάρχει και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ πως είναι η καλύτερη επιλογή. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, να επιστιάσουμε στα όσα μας λέει η νομική επιτροπή, ότι τουλάχιστον στην αρχή δεν μπορούμε να μοιράσουμε την, την ευθύνη με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Αν και προφανώς η απόφασή μας, όπως πάντα, μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα κάνουμε ώστε να αποφύγουμε τις κατηγορίες ότι ότι ίσως να μην είναι τελείως αντικειμενικό. Και σε όλα αυτά, όπως είπα, δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος με την Επιτροπή Σοφών, αλλά σε αυτή την υπόθεση μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι σαφές πως αυτή την συμβεστική ότι αυτή η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη, τα τρία θεσμικά όργανα θα ορίζουν έναν ο καθένας, είναι σαφές για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Μετά το θέμα είναι πώς θα αποπολιτικοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Και εκεί θέλουμε να ακολουθήσουμε την νομική υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε τώρα αυτό το θέμα, σε αυτό το ερώτημα. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει και αργότερα τι θέλει να κάνει τελικά και μέσω του εσωτερικού του κανονισμού. Παράλληλα το σκεφτόμαστε βέβαια. Αλλά δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο τώρα πρέπει να απαντηθεί. Και πάλι είναι μια υποσημείωση δική μου ότι θα είναι δύσκολο να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο εδώ ώστε να αποπολιτικοποιηθεί τελείως το θέμα. Ε, και θα πρέπει όντως να ακολουθήσουμε τη συμβουλή της Επιτροπής ε, ε, της Νομικής Υπηρεσίας να το, να το κρατήσουμε χωριστά. Λοιπόν, πιστεύω πως πάνω κάτω ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να λάβει και την απόφαση. Έχουμε κάπως αποπολιτικοποιήσει το θέμα γιατί ξέρουμε πώς θα εκλεγούν οι, οι, οι σοφοί και αργότερα θα θεσπίσουμε ξεκάθαρους κανόνες όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση και μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο τέλος και αυτό είναι νομίζω σαφές γιατί αυτό μπορεί να προχωρήσει και τη συζήτησή μας. Όπως είπα, νομίζω πως θα συζητήσαμε τα υπόλοιπα θέματα πολλές φορές. Θα πρέπει να εστιάσουμε στα θέματα που είναι καινούργια και είναι καινούργια όσον αφορά την ισορροπία των φύλων. Μα ανέκαθεν ναι, να χρησιμοποιούσαμε αυτή την ισορροπία σε αυτή την Επιτροπή. Όταν λέμε για ισορροπία των φύλων, ξέρουμε τι θα πει. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε και να παίξουμε με τη δικαιοσύνη των φίλων, gender justice κτλ, δεν νομίζω πως θα κερδίσουμε πολλά. Στη χώρα μας αυτό σημαίνει ένα άντρα σε μια γυναίκα και μια γυναίκα. Όταν πρόκειται για το δικό μα πολιτικό κόμμα, α πούμε, στι εκλογικού καταλόγου. Αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε με τόσε λεπτομέρειε. Τι ακριβώ θέλουμε να γίνεται. Όπως είπα, ήδη το έχουμε χρησιμοποιήσει την ισορροπία των φύλων και ξέρουμε περί τίνο πρόκειται. Ας εστιάσουμε λοιπόν στις τελικές τελειοποιήσεις ε, με τις ομάδες μας και να περάσουμε σε μια τελική ψηφοφορία που να μην είναι πολύ περίπλοκη και να γίνει στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ συγκεκριμένα σημεία ήδη συζητήθηκαν, θα προσθέσω και εγώ κάποια, αλλά θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση. Νομίζω ότι η συζήτηση όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη είναι καθοριστική όσον αφορά την εξέλιξη της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει ο καθένας από εμά να κοιτάξει τι συμβαίνει στην χώρα του, σε εθνικό επίπεδο. Ο καθένας από εμά προέρχεται από μια παράδοση και βλέπει πόσο δύσκολο είναι στη δική μας χώρα ο καθένας να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα, να εξελιχθούμε. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη περισσότερη δημοκρατία αν δεν πετύχουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Πρέπει λοιπόν εδώ να φτάσουμε σε κάποιες ε, πιστικές λύσεις. Καταλαβαίνω, όταν κοιτάξει κανείς τη διατύπωση των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών, αυτό είναι μια πάγια πρακτική εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξέβρεση συμβιβασμού. Υπάρχουν διαφορετικές ε, αρχικές θέσεις και προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Και αυτό βεβαίως κάθε φορά που προσπαθούμε να το κάνουμε διαπιστώνουμε ότι η πρώτη μας τάση είναι τελικά να επαναλάβουμε ο καθένας αυτό που θέλαμε αρχικά να πούμε μέσα στην συμβιβαστική τροπολογία. Και το αποτέλεσμα είναι οι εκατοντάδες τροπολογίες. Το αποτέλεσμα πολλές φορές δεν έχει συνοχή βεβαίως. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου εμπειρία και σύμφωνα με τις ε, εμπειρίες που είχα και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο αλλά και εδώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα το συγκεκριμένο απαιτεί έτσι κι αλλιώς συμβιβασμό. Μικρή, μεγάλη, αριστερή, δεξιή θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να έχουμε έναν κανονισμό που να ισχύει για όλους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα έξω. Λυπούμε ιδιαίτερα γιατί μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα. Θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό και είναι και το καθήκον αυτής της Επιτροπής να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό. Βλέπω λοιπόν ακόμα κάποια ανοιχτά θέματα. Παραδείγματο χάρη για το θέμα του πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά την καταγραφή αυτού του συγκεκριμένου καθεστώτος των πολιτικών κομμάτων. Ποιος το κάνει, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να περιγράψουμε αυτή τη διαδικασία με πολύ ακριβή τρόπο. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. η συζήτηση αυτή που έχει οδηγήσει εδώ σε κάποιες ε, συζητήσεις, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις στην Ολομέλεια. Είναι κάτι που ουσιαστικά μας αφορά όλους. Όλοι ανήκουμε σε κάποια κόμματα, όλοι ε, έχουμε κάπου, αν θέλετε, τις ευαισθησίες μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλετε, τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα να μην είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν 100% τις αποφάσεις μας και τις λύσεις που θα προτείνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κάποια άλλα σημεία πιστεύω ότι ακόμα θα πρέπει να προσέξουμε, αλλά αναφέρθηκαν από άλλους συναδέλφους. Το θέμα της κλίδας κατανομής για τη χρηματοδότηση επίσης. Μέχρι σήμερα η συζήτηση συνεχίζεται. Και εδώ υπάρχει σειρά τροπολογιών. Ο συνάδελφος ότι ανέφερε. Εδώ πρέπει να βρεθεί μία συμβιβαστική τροπολογία. Αν γίνεται αυτό, αν κοιτάξει κανείς τις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και καλό θα ήταν αυτό να το κάνουμε πριν την ψηφοφορία να το πετύχουμε πριν ψηφίσουμε. Δεν θα επαναλάβω όλα τα σημεία που ανέφεραν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, με τα οποία συμφωνώ. Σκοπός μας είναι, αν θέλετε, να βρεθεί αυτή η συμφωνία και όντως χρειάζεται χρόνος. Αλλά ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα, περισσότερο χρόνο, επιμονή και υπομονή και να συνεχίσουμε τη συζήτηση έτσι ώστε πραγματικά να μπούμε στην ουσία, να υπάρχει μια ισορροπημένη και σταθμισμένη προσέγγιση. Αλλιώς θα βρεθούμε μπροστά σε μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια η οποία θα είναι δύσκολη, θα είναι δυσάρεστη και αυτό επαναλαμβάνω είναι πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι μία σαφής, ακριβής και καλή ρύθμιση αυτού του θέματος θα είναι προς συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ κύριε Χέφνερ. Μορέιρα. Ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τους όρους για το Μητρό των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, τροπολογία D. Θα ήθελα να στηρίξω τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Γκερέρο. Στο βαθμό που η μεταφορά από την σημερινή σημερινό κομμάτι του άρθρου 13 στο κείμενο που λέτε χάνει την σημασία του ε, το κείμενο που λέει πρέπει να τηρεί ιδιαίτερα στο πρόγραμμά του και στις δραστηριότητές του. Αυτή η φράση έχει χαθεί στην μεταφορά προς το σώμα του 1, έτσι όπως προτείνεται τώρα από την τροπολογία D. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι δεν θα πρέπει να χαθεί. Η παρατήρηση που αφορά το σεβασμό των αρχών ε, της Ένωσης, των ιδιωδών της Ένωσης, το δεύτερο άρθρο πρέπει να διατηρείται τόσο στο πρόγραμμα όσο και στις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Είναι σημαντικό σημείο αυτό. Φυσικά η ισορροπία των φύλων, gender balance τώρα, δεν συνοδεύει και την παρατήρηση του συναδέλφου Σόλτς εγώ πιστεύω πως gender balance είναι μια ε, δόκιμη φράση, αφήνει ένα περιθώριο ε, είναι αντίθετο από το ισότητα των φύλων, ε, είναι διαφορετικό μάλλον, ενώ η ισορροπία των φύλων μπορεί να παίρνει κάποια, κάποιες μεταβλητές. Σημαίνει ότι κανένα από τα δύο φύλλα δεν θα πρέπει να είναι 100% στους εκλογικούς καταλόγους ή δεν θα πρέπει να κατέχει δύο ε, διαδοχικές θέσεις στον κατάλογο. Πιστεύω πως αν αυτό είναι συμβατό με το gender balance, τότε εντάξει ισορροπία λοιπόν των φύλων στα κόμματα, ώστε να υπάρχουν κάποια όρια και να τηρείται η ισορροπία. Τρίτη μου παρατήρηση προκύπτει από τις παρατηρήσεις του συναδέλφου Χέφνερ, γιατί πιστεύω ότι στον έλεγχο, στην επαλήθευση, του κατά πόσο σέβονται τις αρχές της Ένωσης στα πολιτικά κόμματα, δεν θα πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο ώστε να μπορεί κανείς να σκεφτεί πως υπάρχει πολιτική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι εμείς αφισβητούμε την ίδια μας την ύπαρξη, όπως είπε ο συνάδελφος Χαφνερ. Γι' αυτό και η Επιτροπή Σοφών που αναφέρθηκε και υπήρχε στην πρόταση της Κομισιόν είναι καλή κατά τη γνώμη μου αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα, ότι το Κοινοβούλιο δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εκθέσεις της Επιτροπής των Σοφών. Δεν θα πρέπει όμως ε, να πολιτικοποιηθεί αυτό το θέμα. Πιστεύω επίσης ότι αυτή η ιδέα της ανεξάρτητης αξιολόγησης των πολιτικών ιδεών, των αξιών της Ένωσης και είμαστε στο 13ο άρθρο της νομοθετικής πρότασης θα πρέπει να ισχύει για την αξιολόγηση των, στάνταρ των πολιτικών κομμάτων και το gender balance θα έπρεπε να είναι αντικείμενο κάποιας αξιολόγησης ανεξάρτητης, αντί να είναι μόνο αυτή η Επιτροπή η, του Κοινοβουλίου, η πολιτική που εκτιμά κατά πόσο διοργανώνονται τα κόμματα με βάση τις ε, δημοκρατικές προδιαγραφές. Θα έπρεπε λοιπόν να εφαρμόσουμε και να πετήσουμε την αξιολόγηση και την επαλήθευση των δημοκρατικών προδιαγραφών και τη στήρισή τους με βάση αυτές τις έννοιες που βρίσκονται στο άρθρο 4 στη δεύτερη παράγραφο της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ό,τι και αν κάνουμε για να απομακρύνουμε οποιαδήποτε ιδέα πολιτικής αυθαιρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επαλήθευση των πολιτικών ενιών ή αντιλήψεων είναι θετικό. Ε, θα πρέπει να μειώσουμε το περιθώριο διακριτικής και να εκμεταλλευτούμε την ύπαρξη της Επιτροπής των Σοφών για να επαληθεύσει και την δημοκρατική οργάνωση και την ισορροπία των φύλων όπως, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 της παρα, ε, εδάφιο 2. Και όσον αφορά τις συμβιβαστικές τις εισηγήτριες είναι λογικές, ισορροπημένες και αξίζουν να υποστηριχτούν από την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Γιαννάκου, αν θέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν θέλω να σημειώσω ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη την εμπειρία με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αν και αυτά έχουν ένα στάτους μη κυβερνητικής οργάνωσης. Δεν είναι δηλαδή ευνίδιο, ούτε πέφτουμε από τον ουρανό. Έχουμε ήδη μία συγκεκριμένη εμπειρία. Και δεν έχουμε φαινόμενα μέχρι σήμερα να σε κανείς το μέσο αυτό για να εκδιώξει ή να εκβάλει ένα πολιτικό κόμμα. Νομίζω ότι η φόβη αυτή είναι υπερβολική. Τώρα θα απαντήσω συγκεκριμένα επί όσων παρατηρήσεων έγιναν, αφού σημειώσω κύριε Πρόεδρε ότι από 13 Μαρτίου έχουν όλοι τις τροπολογίες τις συμβαστικές και κανείς δεν μου έχει στείλει καμία παρατήρηση. Για να είμαστε ειλικρινείς και να μην παριστάνουμε ότι δεν ξέρουμε εδώ πέρα. Δεν έχω πάρει από κανέναν παρατηρήσει. Ο κύριος Νταφ μιλάει για το σημείο 5, για την νομική προσωπικότητα. Η νομική προσωπικότητα δημιουργείται μέσω αυτού του κανονισμού. Ό,τι δεν ρυθμίζεται μέσω αυτού του κανονισμού ρυθμίζεται από τα κράτη-μέλη στα οποία θα είναι εγκατεστημένο το κόμμα. Εάν παραδείγματο χάρη ένα πολιτικό κόμμα εγκατασταθεί στο Λονδίνο, ό,τι δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό θα ρυθμιστεί με βάση τους νόμους και τους κανόνες για τα πολιτικά κόμματα στη Βρετανία. Επομένως έχουμε αυτόνομη νομική προσωπικότητα. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να μπούμε σε απίθανες λεπτομέρειες διότι και το κράτος μέλος στο οποίο θα είναι εγκατεστημένα τα κόμματα έχει δικαίωμα σε ορισμένα ζητήματα και πληροφορίες να δώσει και να συνεργαστεί και να ελέγξει εκεί που δεν ελέγχει αυτός ο κανονισμός. Η οργάνωση του Κοινοβουλίου προϋπάρχει. Όπως ξέρουμε έχουμε τον, τον εσωτερικό μας κανονισμό. Ήδη στην υπάρχουσα κατάσταση προβλέπονται τα τρία πρόσωπα, τα τρία, οι τρεις σοφοί οι οποίοι θα κρίνουν τα πολιτικά κόμματα. Και εν συνεχεία ακολουθείται ο κανονισμός του Κοινοβουλίου. Τώρα εκεί μπορούμε, όπως σωστά είπε ο κύριος Τσαρκόφσκι, εν συνεχεία και αφού εγκριθεί αυτό, να δούμε αν χρειάζονται μέσα στον κανονισμό του Κοινοβουλίου ορισμένες τροποποίησεις δεν μας εμποδίζει κανένας κύριε Πρόεδρε να το κάνουμε αυτό. Σημείωσε την παραβίωση των αρχών της Ένωσης ο κύριος Ντάφ. Πράγματι όλοι ανησυχούμε και μάλιστα ορισμένα κόμματα ανησυχούν διότι υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν είναι υπέρ της ύπαρξης της Ένωσης. Και αναρωτιούνται θα υπάρξει θέμα για αυτούς. Το αντικείμενο δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ακριβώς το σημείο σε το οποίο σημείωσε ο κύριος Γκερέρο και ο κύριος Μορέιρα στο οποίο δεν έχω αντίρρηση να μείνει κύριοι συνάδελφοι. Ας μείνει δύο φορές. Δεν πειράζει. Ας μείνει και εκεί διότι οι αρχές αυτές πράγματι είναι οικουμενικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών είναι παγκόσμιες αρχές επομένως οι παραβιάσεις αφορούν σε παραβίαση αρχών και αξιών που είναι και παγκόσμιες αρχές και αξίες όχι στο αν είναι υπέρ της εξέλιξης της Ένωσης ή όχι. Επομένως δεν υπάρχει φόβος για κάποια κόμματα που υπάρχουν ήδη στο Κοινοβούλιο και που δεν ε, αποδέχονται ε, ορισμένα, ορισμένες ε, εξελίξεις που αποδέχονται άλλα μέλη του Κοινοβουλίου και άλλα κόμματα. ο κύριος Μπρόντ σημείωσε το σημείο Α και είπε υπενισόμεθα ότι αυτά τα κόμματα θα είναι excluded που δεν θα είναι εγκεκριμένα από την καθεστική απολυτική τάξη. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Κανείς δεν έχει εμποδίσει να εμφανιστούν κόμματα και να είστε βέβαιοι ότι στις επόμενες εκλογές θα εμφανιστούν κόμματα που δεν έχουν καμία σχέση με την καθεστική απολυτική τάξη. Ήδη εμφανίζονται σε όλες τις χώρες. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να θέσει αυτό τον υπενιγμό ως θέμα διότι δεν έχει τεθεί και μέχρι σήμερα. Δεν έχει τεθεί για τα υπάρχοντα κόμματα μέχρι σήμερα. Τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ο κύριος Σόλτς. Θα επανέλθω σε αυτά που είπε και ο κύριος Τσαρκόφσκι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε για να προσβάλλει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου αλλά η διαδικασία ελέγχου πρέπει να γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προσφυγή στο δικαστήριο μπορεί να γίνει όπως περιγράφεται στις συνθήκες. Δεν μπορεί κάθε αίτημα ή κάθε παράπονο να πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γελιοποιήσει το θεσμό. Αλλά το δικαστήριο είναι πάντα εκεί. Και γνωρίζοντας η πολιτική τάξη όπως την αναφέρατε ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μπορούν να προσληθούν οι αποφάσεις, νομίζω ότι αυτό και μόνο καθιστά πάρα πολύ προσεκτικό το Κοινοβούλιο σε όλες τις εκφράσεις του. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έθεσε ο κύριος Σόλτς προφανώς εννοείται το 85-15 που γίνεται στη δική μου πρόταση 90-10. Ε, νομίζω ότι είναι πιο δημοκρατικό είναι δηλαδή πιο δημοκρατικό να δώσουμε κάτι παραπάνω στα κόμματα με βάση την αποδοχή που έχουν από τους πολίτες. Και εν συνεχεία κατά ισότιμο τρόπο το 10%. Τώρα το gender balance. Κύριοι συνάδελφοι βάλαμε τον όρο gender balance διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα κόμμα επειδή δεν έχει 50% και 50% ε, μέλη στο, στα διάφορα όργανα του κόμματος. Ούτε μπορούμε να αποκλείσουμε αύριο να γίνει ένα κόμμα μόνο από γυναίκες παραδείγματο χάρη. Δηλαδή δεν μπορούμε να το γράψουμε αυτό. Το gender balance υπενήσεται ευθέω, μάλλον όχι υπενήσεται, τονίζει ευθέω τις ίσες ευκαιρίες. Λέμε ισορροπία και των δύο φύλων. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Και η έννοια του promotion. Γιατί αλλιώς εγώ δεν ξέρω κανένα κόμμα στην Ευρώπη που μπορεί να εξασφαλίσει ότι μέσα στα όργανα του είναι 50% γυναίκες. κανένα πραγματικά δεν ξέρω. Ούτε εσείς έχετε κόμματα, κανένας. Στα κόμματά σας δεν έχει κάτι τέτοιο που μπορεί και δεν μπορεί να επιβληθεί δημοκρατικά. Διότι δεν μπορεί να επιβληθεί στους πολίτες η συμμετοχή. Ευκαιρίες μπορούν να δοθούν. Ε, για το ΣΕ είπα ότι εντάξει συμφωνώ κύριε Γκερέρο να διατηρηθεί. Δεν πειράζει, ας είναι δύο φορές. Γιατί εδώ στο σημείο ΣΕ πράγματι έχει αναλυτικότερα τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό των μειονοτήτων κτλ. Οπότε εκεί συμφωνώ. Ε, τώρα, η Επιτροπή Σοφών, κοιτάξτε, υποθέτω ότι τα τρία όργανα θα ορίσουν κάποιες προσωπικότητες ε, που θα μπορούν να δουν τα πράγματα με αντικειμενικότητα και από απόσταση. Νομίζω ότι σε κάποια περίπτωση που είχε τεθεί θέμα είχε ε, υποδηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας ανησυχεί. Εν τω μεταξύ το Κοινοβούλιο όμως έχει όλη τη δυνατότητα να καλέσει αυτούς που εκφράζουν παράπονα, να κάνει ένα hearing κτλ, να εξετάσει ένα θέμα. Ε, ο κύριος Χέφνερ μίλησε για εκατοντάδε τροπολογίε χωρί συνοχή. Ε, δεν φταίω εγώ που γίνονται εκατοντάδε τροπολογίε χωρί συνοχή, κύριε Χέφνα. Αυτοί που τι κάνανε φταίνε. Δεύτερον, λέτε ότι απαιτείται συμβασμό. Ναι, βεβαίω απαιτείται συμβασμό. Αλλά δεν είναι, ε, δεν είναι πάντοτε επιτεύξιμο ένα συμβιβασμό. Δεν έχουμε όλοι τι ίδιε απόψει. Γενικά, αναφέρατε ορισμένα πράγματα ότι ε, ε, ε, το θέμα της χρηματοδότησης ότι δεν είναι σαφής ο κανονισμός ακριβής και δεν υπάρχει καλή ρύθμιση κλπ. Είπατε όμως γενικότητες κύριε Χέφνερ. Είχατε την ευκαιρία από τις 13 Μαρτίου να μου στείλετε συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Δεν είπατε τίποτα συγκεκριμένο. Τίποτα απολύτως συγκεκριμένο δεν είπατε. Τέλος ο κύριος Μορέιρα εζήτησε να παραμείνει η τροπολογία την οποία ανέφερε ο κύριος Γκερέρο, η τροπολογία C και νομίζω ναι τελικά αυτό είναι σωστό γιατί όπως είπα πριν εκφράζει τις γενικότερες απόψεις. Κύριε Πρόεδρε θέλω να μου επιτρέψετε να επανέλθω στη Λίγκα να σας θυμίσω τι δεν αποδεχόμαστε από τη Λίγκα του Κοινοβουλίου με βάση τις προτάσεις που έχουν γίνει από τα μέλη δεν αποδεχόμαστε ότι μόνο κόμματα θα μπορούν να φτιάχνουν ευρωπαϊκό κόμμα και εκλεγμένοι βουλευτές και ευρωβουλευτές. Έτσι διευρύνουμε το πεδίο, συμφωνώντας με την άποψη της Επιτροπής. Διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Αυτό είναι πιο δημοκρατικό. Δεύτερον, η διαδικασία ελέγχου, όπως είπα πριν, μπορεί να καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο τρόπος που το Κοινοβούλιο θα ρυθμίσει την εγγραφή και τον έλεγχο μπορεί κάλλιστα να ρυθμιστεί από τις εσωτερικές διαδικασίες και τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου. Αυτό υπάρχει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η γνωμοδότηση δίνει σημαντικό ρόλο στην ανεξάρτητη επιτροπή των τριών επιφανών προσώπων και όπως είπα πριν συμφωνούμε. Και τέλος το κομμάτι, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να μπορούν να συμμετέχουν σε εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και σε δημοψηφίσματα που συνδέονται με την αλλαγή των συνθήκων και τις πολιτικές της Ένωσης είπα να το αφήσουμε για τον τρίλογο γιατί υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου η εμπλοκή ευρωπαϊκών κομμάτων στα δημοψηφίσματα συναντά νομικές δυσκολίες, συνταγματικές μάλλον δυσκολίες. Επομένως αυτό το κομμάτι μπορούμε να το αφήσουμε στον Τρίλογο. Κατά συνέπεια, καταλήγοντας κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα ε, από εδώ και πέρα να κάνουμε μια συνάντηση πάλι με τους Σάντους για να συγκεκριμενοποιηθεί και η άποψη των ε, σκιωδών εισηγητών για τις τροπολογίες που δεν είναι συμβιβαστικές και είναι αρκετές και να μπορούμε να προχωρήσουμε στο Στρασβούργο χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ψήφιση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε τώρα πλέον το συγκεκριμένο θέμα, επιβεβαιώνοντας αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή ότι θα υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση στις 15 Απριλίου στο Στρασβούργο. Στην ημερήσια διάταξη θα είναι μόνο το συγκεκριμένο θέμα και ε, θα αποφασίσουμε να συνεχίσουμε ε, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση μόνο στην ψηφοφορία. Ταυτόχρονα η εισηγήτριά μας ε, θα έρθει σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές και θα προσπαθήσει να μας ε, ε, διευκρινίσει με σωστότερο τρόπο ε, τα προβλήματα τα οποία σημειώθηκαν από τους συναδέλφους. Για να κλείσουμε ένα πράγματι πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, για το 12. Πήραμε ήδη την αδειοδότηση της διάσκεψης των Προέδρων για μία έκθεση πρωτοβουλίας. Όπως είπαμε ορίστηκαν δύο εισηγητές, οι κύριοι κύριοι Φόξ και και ε, σήμερα βάλαμε το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ακούγοντας τους πρώτα βέβαια, να μας πούν ποιες είναι οι πρώτες τους ιδέες. Ο κύριος Φόξ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γέδρες και ο καθορισμός μάλλον των εδρών των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά επρόκειτο για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχικά τουλάχιστον αυτό ήταν το θέμα. Και φυσικά θα υπάρξει ε, εστιασμός στο θέμα αυτό. Είναι κάτι που βεβαίως ε, είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει το πρωτόκολλο 6 της συνθήκης που καθορίζει το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει μια πρόταση τροπολογίας αυτού του πρωτοκόλου και από εκεί και πέρα χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Υπάρχει η μεγάλη πλειοψηφία συναδέλφων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καταρχήν είναι υπέρ της μίας και μοναδικής έδρας και αυτό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κάποιοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Κάποιοι θεωρούν ότι μολύνουμε το περιβάλλον μεταφέροντας κάθε μήνα όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την μία έδρα στην άλλη, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι το επιδικόμενο για ένα φιλικά προς το περιβάλλον κοινοβούλιο. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ε, για άλλους λόγους επιθυμούν να υπάρχει μία και μοναδική έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποιοι και να είναι πάντως οι λόγοι, χρειάζεται μία ολοκληρωμένη συζήτηση για το θέμα αυτό. Και εκπλήσωμαι γιατί τα τέσσερα χρόνια της δικής μου θητείας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποτέ δεν προέκυψε αυτό το θέμα. Και εγώ όταν εξηγώ στην εκλογική μου περιφέρεια ορισμένα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ερωτήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την διπλή έδρα προκύπτουν συνεχώς και σε πολλές περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν είναι πρόθεσή μου εδώ τώρα και ελπίζω να μην μπούμε ε, σε αυτήν την συζήτηση για το ποια θα είναι η έδρα που θα πρέπει να επιλέξουμε εάν ε, τελικά θα επιλεγεί μία έργα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πραγματικά να περιοριστούμε στην ουσία. Ο κύριος Αφνερ και εγώ ουσιαστικά έχουμε προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα, θα σας το μοιράσουμε, με αρκετό χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε εις βάθος το θέμα. Αυτό και να ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Θέλουμε λοιπόν μια πλήρη και εις βάθος συζήτηση και βεβαίως θα πρέπει να εμπλακούν και να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή και οι κυβερνήσεις οι οποίες ε, εμπλέκονται καθότι μία από αυτές τις έδρες είναι ε, στην χώρα τους. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε λοιπόν με την γαλλική, την βελγική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, με έναν τρόπο που να ε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη και με μεγάλο σεβασμό τις δικές τους παρατηρήσεις και ε, απαιτήσει και ο κύριος Άγνιου, ο συναδελφός μου, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πώς εκφράζεται. Ξέρω ότι καμιά φορά μιλάμε εδώ σκεπτόμενοι πώς θα εντυπωσιάσουμε τους ψηφοφόρους μας. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείξουμε σεβασμό προς τους άλλους συναδέλφους και το λέω αυτό προς όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Προσέξτε το λεξιλόγιό σας. Αν ακούσετε ένα έντονο ή αγενές τρόπο έκφρασης από κάποιο συνάδελφο από τη Μεγάλη Βρετανία, και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφραστεί αν ναι ή όχι θέλουμε μία έδρα. Εγώ ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα τροποποιηθεί το πρωτόκολλο 6 και ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει συζήτηση στο Συμβούλιο. Σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας δίνουμε μια πρώτη ευκαιρία να ακουστούν οι άλλοι σκιώδεις και οι άλλες πολιτικές ομάδες. Αποφασίσαμε να αρχίσει τη συζήτηση και εγώ να την ολοκληρώσω. Οπότε, για να έχουμε αρκετό χρόνο και για τους συναδέλφους, δεν θα πρέπει να μακρηγορήσω τώρα, αλλά να θέσω και πάλι τα ερωτήματα, γιατί είμαστε στην αρχή της έκθεσης. Έχουμε φτιάξει ένα ένα σκελετό για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Θα σας το, διανέμουμε τώρα και σήμερα θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις για να μπορέσουμε να τις λάβουμε υπόψη από την πρώτη στιγμή στη σύνταξη της έκθεσης και θέλουμε να συνεργαστούμε με όλα τα μέλη όλων των ομάδων. Ωραία, ευχαριστώ. Το σκελετός, όπως είπα, το πρόγραμμα έχει διανεμηθεί και τώρα ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Αγνιού. Πρόεδρε, με κολλάκεψε πολύ η εισαγωγή του κυρίου Φόξ. Δεν ξέρω αν εγώ θα τον απογοητεύσω, θα δούμε. Αλλά όταν μιλάμε για την τοποθεσία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, βασικά μιλάμε για αυτό το παραλογισμό του να έχουμε δύο έδρε για, για το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ε, δυνατότητα κατά ε, τοποθέτησης μια υπηρεσία ενό οργανισμού, ε, όμως είναι σπάνιο να έρθει καμία στη δική σου χώρα. Πρόσφατα Ε, έγινε λόγος ε, για έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ευρεσιτεχνίες στο Λονδίνο, αλλά φαίνεται πως ε, τελικά δεν είναι πολύ εύκολο ε, το πράγμα. Αυτό το οποίο πραγματικά εξοργίζει τους ε, δικούς μου εκλογείς είναι η εκείνη υπόθεση όπου ε, κάθε μήνα χρειάζεται χιλιάδες άνθρωποι να ταξιδεύουν πέρα σε μια επαρχιακή γαλλική πόλη, να ζουν με μια βαλίτσα παραμάσχαλα και μετά να πρέπει στο τέλος της εβδομάδας να ξαναγυρνάνε πίσω χιλιάδες χιλιάδων ε, και εκατομμύρια ευρώ χάνονται και όλα αυτά υπέρ της ματοδοξίας ε, των ε, Γάλλων και για να επιβιώνει η οικονομία του Στρασβούργου. δαπανώνται ένα σωρό χρήματα λοιπόν χωρίς λόγο τη στιγμή που 50% των νέων της Ελλάδας ε, έχει μείνει άνεργο. Ξέρω πως υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να ακούει για την ε, Ελλάδα, αλλά στη χώρα μου η διάσωση της Ελλάδας κόστησε τη δεύτερη φορά 10 δις λίρες ε, και ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί. Ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να συμφωνήσει και στην Κύπρο ακόμα 10% θα φορολογήσουν ε, από τις αποταμιεύσεις ε, των ε, καημένων των Κυπρίων. Λοιπόν, ας δοθεί επιτέλους μια τιμιγορία για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λεγκρίπα. Λεγκρίπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που μια επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμως βάζει στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της το θέμα του καθορισμού των εδρών των θεσμικών οργάνων. Αυτός είναι ο τίτλος του εγγράφου της έκθεσης, όπως καθορίστηκε από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων και βεβαίως Όλοι εδώ θα βασιστούμε στην σοφία, στον αμοιβαίο σεβασμό που επικρατεί εδώ στην ε, Επιτροπή μας ε, συνήθως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και θα πρέπει να συζητηθεί στο σωστό επίπεδο. Μιλούμε για τις έδρες ε, των θεσμικών οργάνων. Όπως σας είπα, αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης αυτής, αλλά όπως είπαν και οι δύο συνεισηγητές, δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Αυτό που κυρίως θα μας απασχολήσει, αυτό που κυρίως θα συζητήσουμε, είναι ο καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφασίσει για την έδρα του, για το πού θα είναι η έδρα του. Γι' αυτό και θα πρέπει εδώ Αν κοιτάξω πολύ προσεκτικά το χρονοδιάγραμμα που μας προτείνουν σήμερα οι συγητές, που προβλέπει αρκετό χρόνο, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία έδρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρωτόκολλο 6 καθορίζει το Στρασβούργο σαν την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλοί τόποι εργασίας, αλλά όταν αναφέρεστε στην καμπάνια για την μία και μοναδική έδρα, one single seat, αυτό ουσιαστικά υπάρχει ήδη. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία, μία και μοναδική έργα, το Στασβούργο. Αυτό λοιπόν ήδη υπάρχει. Αυτό το αναφέρω καθαρά όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Πρωτόκολλο 6, άρθρο 341 για τον καθορισμό της έδρας και η απόφαση του Συμβουλίου του 92 στο Εδιμβούργο, η συνθήκη του Άμστερνταμ, όλα αυτά επιβεβαιώνουν καθώς και η συνθήκη για τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι αποφάσεις, οι πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου, η τελευταία του Δεκεμβρίου. Σκοπός μας λοιπόν εδώ είναι να επιλέξουμε αν η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επαναλαμβάνω έχει επιλεγεί για το Στρασβούργο, μια σημαντική πόλη για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, μια πόλη που εμπεριέχει το DNA της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της ειρήνης, γι' αυτό και τελικά ε, επελέγει η πόλη του Στρασβούργου σαν μια πόλη που εκφράζει το πνεύμα της συμφιλίωσης και της ειρήνης. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα, σε μια δύσκολη, ταραγμένη εποχή για την Ευρώπη, η μνήμη είναι κάτι που θα πρέπει να μας εμπνεύσει. Είναι τμήμα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια ιστορική συνεισφορά για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε έτσι ώστε να μην υπάρξει εδώ καμία αλλίωση της μνήμης και να μην ξεχάσουμε τις βασικές αξίες οι οποίες ε, θεμελίωσαν την ίδρυση της ε, Ευρώπης. Οι πατέρες της Ευρώπης και οι πρώτες χώρες που ξεκίνησαν ε, την Ευρώπη επέλεξαν την πόλη του Στρασβούργου για όλους αυτούς τους λόγους. Τώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί χώροι εξουσίας και πολλοί χώροι εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια έδρα, αλλά πολλοί χώροι εργασίας, τόποι εργασίας, το Λουξεμβούργο, οι Βρυξέλλες, που είναι κυρίως η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλές άλλες πόλεις και τόποι εξουσίας με άλλους θεσμούς, υπηρεσίες, κέντρα αποφάσεων. Αυτό δείχνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι πραγματικά είμαστε ενωμένοι μέσα σε ένα πνεύμα πολυμορφίας και διαφορετικότητας. Και αυτό ξεκίνησε από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το πνεύμα που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση η πολυμορφία, η πολυεθνικότητα, η κινητικότητα. Μα αυτό είναι ουσιαστικό για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η κινητικότητα. Και αυτό βεβαίως σε όλη την ευρωπαϊκή ε, επικράτεια. Οι πολιτικοί της Ευρώπης δείχνουν με αυτήν την ε, κινητικότητά τους ότι εμπνέονται από το ευρωπαϊκό πνεύμα. Και βεβαίως η ιδέα του να συγκεντρωθούν όλοι οι χώροι εξουσίας. Γιατί τελικά αυτό είναι το μήνυμα αυτών που προωθούν αυτή την συγκέντρωση όλων των θεσμικών οργάνων και όλων των ε, τόπων εργασίας και την μεταφορά τελικά της έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου στις Βρυξέλλες είναι για μένα παράδοξο γιατί αυτό βέβαια μας οδηγεί στη συζήτηση επί της ουσίας, αλλά με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε, αν θέλετε, τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής πρωτεύουσας, μιας ευρωπαϊκής Washington DC. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα παράδοξο ε, φαινόμενο, γιατί αυτοί που το προτείνουν δεν είναι καθόλου οι υπέρμαχοι μιας ομοσπονδίας. Θέλουν παρόλα αυτά να συγκεντρώσουν σε μία μοναδική πρωτεύουσα όλες τις εξουσίες, την εκτελεστική, την νομοθετική, όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν εδώ ότι η αρχή της κινητικότητας, η αρχή της πολυμορφίας, η αρχή του πολυκεντρισμού είναι κάτι που θα πρέπει να μας οδηγήσει αντίθετα στο να κατανείμουμε κέντρα αποφάσεων, κέντρα εξουσίας σε πολλούς τόπους, σε πολλές πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πραγματικά χαρακτηρίζει τις προσπάθειές μας, που δεν είναι πάντα εύκολες. Επαναλαμβάνω, στη δύσκολη εποχή που ζούμε, στις προσπάθειές μας να πλησιάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να μειώσουμε την απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών. Και νομίζω ότι η υπερσυγκέντρωση σε ένα ενιαίο και μοναδικό χώρο, σε μια πόλη, είναι κάτι που δεν θα μας διευκολύνει. Θα αυξηθούν αντίθετα οι επικρίσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι λοιπόν κατά την απόψή μου σημαντικό η άποψη, η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών, των οποίων είμαστε εκφραστές, η νομοθετική εξουσία, την οποία εκφράζουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ακουστεί, να εκφραστεί και να μπορεί να ακουστεί κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη από αυτή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ του να διατηρηθεί στην Ευρώπη ένα σύστημα πολυκεντρικό, με πολλά κέντρα εξουσίας. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση απλώς ξεκινάει και δεν πιστεύω ότι η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια εδώ αυτή τη στιγμή για να εκφραστεί όσον αφορά τα θέματα κόστους. Ίσως κάποια στιγμή να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά και να διορθώσουμε κάποιους αριθμούς που κυκλοφορούν οι οποίοι δεν είναι πάντα ορθοί. Εν πάση περιπτώσει θα οργανωθεί και μια ακρόαση ενδεχομένως το Μάιο και καλό θα ήταν να δούμε την ομιμότητα και την ορθότητα μιας επιλογής γιατί πιστεύω ότι δεν συμφωνούν όλοι, <clears throat> όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι εθνικές αρχές, ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει αυθόρμητα και από μόνο του για το πού θα είναι η έδρα του. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και τα πολιτικά μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε στους ψηφοφόρους μας και αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Γετεμάκη. puhun suomea. Edellinen puheenvuoro oli hyvin ymmärrettävä ja minun täytyy sanoa, että silloin kun Euroopan... Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ήταν το θέμα που συζητάμε είναι σωστό να το συζητήσουμε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποφασίστηκε η έδρα του Κοινοβουλίου ναι, είναι στο Στρασβούργο. Ήταν πολύ σωστό τότε. Υπήρχαν έξι κράτη-μέλη, αν δεν κάνω λάθος. Και η επιλογή της συγκεκριμένης έδρας και της συγκεκριμένης πόλης είχε καθοριστεί από, θα έλεγα, τον μεγάλο αυτό πόλεμο που είχε προηγήθει. Και γι' αυτό η απόφαση που είχε ληφθεί τότε ήταν μια σοφή και σωστή απόφαση. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να φέρουμε στους ώμους μας το βάρος της ιστορίας. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενηλικιωθεί, να ζήσει στο παρόν, να ζήσει στο μέλλον με αποτελεσματικό τρόπο και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το πολιτικό μήνυμα που θα στείλουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα το οποίο τώρα στέλνουμε στην παρούσα φάση είναι ότι σκοτιστήκαμε για το κόστος. Ε, ξοδεύουμε δεξιά και αριστερά τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Πράγματι έχουμε ένα τεράστιο λογαριασμό να πληρώσουμε ε, κάθε χρόνο για το Στρασβούργο, αυξάνουμε συνεχώς φυσικά το ίχνος του διοξιδίου άνθρακα το οποίο παράγουμε, δεν το έχουμε μειώσει καθόλου και δεν δείχνουμε να ανησυχούμε ε, που δεν το έχουμε μειώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα στους πολίτες μας. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να το στέλνουμε. Ε, όχι βέβαια. Και θα πρέπει να ε, μιλήσουμε λίγο και για την αποτελεσματικότητα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς απαιτούμε από όλους γύρω μας να εργαστούν σκληρά, να εργαστούν ευθυνά, να εργαστούν ανταγωνιστικά. Και εμείς πώς εργαζόμαστε. Δεν είμαστε αποτελεσματικοί, φυσικά, το τσίρκο αυτό το οποίο περιοδεύει τακτικά στην πόλη του Στρασβούργου ε, σε τις άλλη ε, δυσκολεύεται και να το κάνει γιατί εγώ ας πούμε για να πάω στο Στρασβούργο πρέπει να ξυπνάω στις 5 η ώρα το πρωί για να τα καταφέρω και δεν είναι ε, καθόλου μα καθόλου εύκολο για να επιστρέψω αναγκάζομαι να να ταξιδεύω μέχρι τα μεσάνυχτα πάλι. Αναγκαζόμαστε για να τα συμπτύξουμε όλα, να εργαζόμαστε καθόλου αποδοτικά τη νύχτα της Τρίτης, τη νύχτα της Τετάρτης και είδαμε και μάλιστα την προηγούμενη Τετάρτη πόσο επικίνδυνη στην ανθρώπινη υγεία είναι αυτή η συνεχής αγχώδης μετακίνηση. Και κατανοώ δυστυχώς πολύ καλά γιατί ο αγαπητός μας αντιπρόεδρος, ο κύριος Παπαστάμκος, υπέστη αυτό το τόσο σοβαρό επεισόδιο. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ανθρώπινος ο τρόπος αυτός. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο να συμπτήσουμε το μήκος, τον χρόνο μάλλον των εργασιών μας με καταστροφικά αποτελέσματα όπως δυστυχώς βιώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πρέπει να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πια ότι έχουμε μία έδρα. Όλος ο κόσμος δουλεύει στο ίδιο σημείο, στον ίδιο χώρο, στην ίδια πόλη, με αποτελεσματικό για την Ευρώπη τρόπο, με αποτελεσματικό για τους πολίτες της Ευρώπης τρόπο. Δεν μπορώ πια να καταλάβω καθόλου το πώς κάποιοι σήμερα συνεχίζουν να πιστεύουν ότι να πηγαίνουμε στο Στρασβούργο ε, κάθε μήνα είναι μια καλή ιδέα. Εντάξει, κάποτε ήταν μια καλή ιδέα, αλλά άνθρωποι είμαστε, αλλάζουμε αποφάσεις. Γιατί αν δεν αλλάζαμε ποτέ αποφάσεις θα είχαμε καταδικαστεί στην αναποτελεσματικότητα. Επαναλαμβάνω, όταν ελήφθη η απόφαση για το Στρασβούργο ήταν μια σωστή απόφαση. Τώρα είμαστε 27 χώρες. Έχουμε εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας. Έχουμε διαφορετικές αρμοδιότητες. Δεν είμαι θα μια απλή λέσχη συζητήσεων τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδρίαζε κάπου κάπου, δεν ονομαζόταν καν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ τώρα συνεδριάζει ε, θεσμικά, συνεδριάζει τακτικά και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την διατήρηση του Στρασβούργου σαν έδρας του Κοινοβουλίου. Η ακρόαση λοιπόν είναι μια καλή ιδέα, επιτέλους να γίνει αυτή η συζήτηση και θα ήθελα να καλέσουμε και προσκεκλημένους ε, εκπροσώπους των κρατών μελών να μας πούν επιτέλους και τα κράτη-μέλη τι πιστεύουν γι' αυτό. Γιατί ο μοναδικός τρόπος ε, για να καταλάβουμε τι θέλουν τα κράτη-μέλη είναι να τους θέσουμε ερωτήματα. Ευχαριστώ κυρία Γιάτεμάκη. Ο κύριος Γουαλτιέρη. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα ξεκινάμε μια συζήτηση που είναι πολύ σημαντική και που είναι και λεπτή θέμα. Θα πρέπει με πολύ σοβαρό τρόπο να το συζητήσουμε και γι' αυτό πρέπει να πω πως εκτίμησα την εισήγηση του συναδέλφου Φόξ. Πιστεύω πως τα πρώτα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε σήμερα αφορούν το χρονοδιάγραμμα και τον χαρακτήρα αυτής της έκθεσης. Για το χρονοδιάγραμμα έχουμε εδώ μια πρόταση προγράμματος. Διερωτώ με μήπως η απέτηση να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εις βάθος αυτήν την έκθεση θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα χρονοδιάγραμμα ελαφρώς πιο σφιχτό, διότι σίγουρα δεν χρειάζεται με βιασύνη να προχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα ίσως και 7-8 μήνες ε, να μπορούσαν κάπως να περιοριστούν. Τώρα, Όσον αφορά το θέμα, τα θέματα μάλλον σίγουρα, κυρίως όσον αφορά τις ε, πιθανές ε, λύσεις, θα είναι σωστό να είμαστε σοβαροί και να κατανοήσουμε πόσο περίπλοκα είναι τα θέματα και ποια είναι η αιτιολόγηση από κάθε πλευρά. Καταρχήν όσον αφορά το νομικό πλαίσιο. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε και να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε με βάση τη γενικότερη τα, τα γενικότερα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ Είμαι ανάμεσα σε εκείνους τους συναδέλφους ε, που είναι κάπως επιφυλακτικοί απέναντι στην ιδέα της μεγαλύτερης ε, ολοκλήρησης και να ξεπεράσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση την αρχή της ε, απόδοσης ή καταχώρησης γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Είναι χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να το ξεπεράσουμε δεν θα είχε νόημα αν περιοριζόταν μόνο σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε ότι ο ορισμός ενός κανόνα των συνθηκών ε, συμβαδίζει με το ευρύτερο πλαίσιο των συνθηκών. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της αρχής competence competence. Άρα είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει εδώ συνοχή. αν θέλουμε να σκεφτούμε πιθανές μεταρρυθμίσεις της συνθήκης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναλύσουμε εις βάθος το νόημα αυτού του πρωτοκόλου στο πλαίσιο το γενικότερο των θεσμικών ε, ε ρυθμίσεων για την Ένωση, σύμφωνα και έπειτα να μετρήσουμε και από το φως της ε, απόφασης με τις επιπτώσεις και το νόημα αυτής και να αντιμετωπίσουμε και το θέμα που δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το πνεύμα, ε, την κατεύθυνση μάλλον των συμπερασμάτων του δικαστηρίου σε σχέση με το όρια του Ευρωκοινοβουλίου και το πρωτόκολλο 6. Και άλλο ένα θέμα έπειτα που θα πρέπει να αναλύσει αυτή η έκθεση και το έθεσε και η συνάδελφος Λεγκρίπ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά καρπός ε, αφηρημένος, ενός αφηρημένου μάλλον νομικού σχεδίου, αλλά είναι απόρρια ιστορικών γεγονότων και δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να το ξεχνάμε να το αποφύγουμε. Ε, το νόημα δηλαδή τόσο από την άποψη ενός ε, μοντέλου όχι υπερκράτους, αλλά ενός πολυκεντρικού μοντέλου σε σχέση με το συγκεκριμένο ιστορικό νόημα που έχει το Στρασβούργο και που θα συνεχίσει να το έχει ως πόλη που εξαιρετικά σημαντική σε σχέση με την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. και να μην λέμε ότι δεν, δεν αγγίζουμε το πρωτόκολλο 6. Τον, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι αποφεύγουμε την έννοια και την αξία της πόλης του Στρασβουργού. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν πρέπει να γίνει, ανεξάρτητα από το αν θεωρεί κανείς πως ε, οι σημερινές ρυθμίσεις θα πρέπει να ξεπεραστούν ή να αλλάξουν. Τέλος, υπάρχει και το θέμα που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ακόμα και δεν είμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, αλλά πιστεύω πως υπάρχουν λειτουργικές εδώ επιπτώσεις και ακούσαμε σίγουρα και κάποιες, ε, ε, κάποια από τα αίτια που αναγκάζουν να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τόσο για να δούμε όντως το προφίλ γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε αξιολογήσεις που διαφορετικά θα προέλθουν από άλλους και δεν θα είναι το ίδιο ακριβή. αλλά και επειδή Γνωρίζουμε πως χρειάζεται να τεθούν όρια στο πόσο κεντρικό είναι αυτό το ζήτημα, γιατί εγώ είμαι κατά της ποσοτικοποίησης του κόστους της δημοκρατίας ως βασικού προβλήματος, γιατί μπορεί κανείς να έτσι να καταλήξει να πει ότι για να κάνουμε οικονομία, Α ε, ας μην κάνουμε εκλογέ φέτος. Η δημοκρατία ξεπερνά οτιδήποτε άλλο, είναι υπερέχει δηλαδή, προηγείται. Οπότε θα πρέπει ναι, να βελτιώσουμε τις διαδικασίες κτλ. να έχουμε δηλαδή ε, και να συζητήσουμε και το θέμα του εισέδρας με σοβαρότητα και γνωρίζοντας ότι μιλάμε για την συμβολική και δημοκρατική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για ένα κόστος οποιοδήποτε. Έπειτα, θα πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι σε διάφορες πτυχές και κάτι τέτοιο θα έδινε και δύναμη σε αυτό το κοινοβούλιο για να προχωρήσει και να προτίσει μια υπέρβαση της σημερινής ε, κατάστασης και εδώ πιστεύω και εδώ αντικαθιστώ τον Σκιώδη Δρούτσα που ε, του είχε κάτι απρόπτω και έπρεπε να, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Είναι κάτι το αναπόφευκτο. Συμφωνώ δηλαδή να τεθεί το θέμα, αλλά ε, πιστεύω ακριβώς που πρέπει να τεθεί με την απαραίτητη σοβαρότητα και την ε, απαραίτητη ε, επίσης κατανόηση των ιστορικών, πολιτικών και νομικών ε, θέσεων που κρύβονται πίσω από το πρωτόκολλο παριθμών 6. Ο κύριος Νταφ. Chairman, um... Table. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα καταρχήν. Λογικό είναι προφανώς. Δεν βιάζουμε ιδιαίτερα, δεν πρέπει να βιαστούμε ιδιαίτερα. Και όπως είπε ο Ρομπέρτο Γκουατιέρη, δεν θα σε καμία περίπτωση να βιαστούμε. Γιατί θα διαπράξουμε σφάλματα. Τα οποία δεν θα μπορούμε μετά να αντιστρέψουμε. Ο κύριος Φόξ έχει δίκιο όταν λέει ότι, όπως είπε και η Κωνσταντς Λεπχή, πρόκειται για προηγούμενο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί για το τι θα αποφασίσουμε. Ακριβώς επειδή πρόκειται για προηγούμενο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την γενικότερη, αν θέλετε, νοοτροπία, τις κοινωνικές πτυχές. Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή που επελέγει το Στρασβούργο. Το Στρασβούργο όπως ε, όλοι γνωρίζουμε είναι μια πόλη στην οποία υπάρχουν πολύ λιγότεροι απόντες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα της παραγωγικότητας, το θέμα της αποτελεσματικότητας και ομολογώ ότι δεν έχω ε, άμεση απάντηση να σας δώσω. Είναι κάτι που θα πρέπει σίγουρα να το επεξεργαστούμε και να το εξετάσουμε με σταθμισμένο και ισορροπημένο τρόπο. Η προσωπική μου, αν θέλετε, ε, επιλογή θα ήταν το Κοινοβούλιο να έχει την έδρα του κοντά κοντά στην κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πού είναι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ερώτημα, το σοβαρό ερώτημα που καλούμεθα να απαντήσουμε. Γιατί η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να είναι απομονωμένη όσον αφορά το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρώπης. Ούτε αυτό λοιπόν εύκολα μπορούμε να το απαντήσουμε. Καθότι το λεγόμενο δεύτερο νομοθετικό σώμα, το οποίο δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τέτοιο, το Συμβούλιο, ίσως θα πρέπει να είναι κοντά μας και βλέπουμε ότι για μας είναι σημαντικό να είμαστε κοντά στα κέντρα εξουσίας, κοντά στους δημοσιογράφους, κοντά σε αυτούς που ασκούν λόμπι για μας τους πολιτικούς. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βεβαίως και άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση ότι θα ακολουθήσει συζήτηση για την τροποποίηση της συνθήκης. Πιστεύω ότι έχω πει ήδη την άποψή μου όσον αφορά με τις συνθήκες της Λισαβόνας και τις πιθανές τροποποίησεις. Έχω εκφραστεί για άλλα θέματα λέγοντας ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ήδη υποστεί πιέσεις που ίσως είναι ανυπόφορες. Και θα πρέπει πολύ σύντομα να ξαναδούμε μια πιο ολοκληρωμένη αναθεώρηση με μια συνέλευση που ενδεχομένως θα πρέπει να ξεκινήσει την άνοιξη του 2015. Αλλά οπωσδήποτε η έκθεση αυτή και άλλες που θα ακολουθήσουν θα μας οδηγήσουν στην απάντηση κάποιων ερωτημάτων που έχουν τεθεί εδώ στην Επιτροπή μας και βεβαίως θα πρέπει να επιλέξουμε σωστά ποια θα είναι η αντιπροσωπεία που θα σταλεί σε αυτήν την συντακτική συνέλευση. Και θα πρέπει επίσης να επιλέξουμε προσεκτικά και τα σημεία που θα βάλουμε στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνέλευσης. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω στους ε, εισηγητές για τον ε, τίτλο αυτής της ε, έκθεσης «Καθορισμός της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι προτίθεστε να κάνετε και να πείτε όσον αφορά τις έδρες των άλλων θεσμικών οργάνων. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό το θέμα. Ο κύριος Μπρόντζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Το θέμα του κόστους είναι καθοριστικό. Πριν γίνω μέλος, ε, μερικούς μήνες, ε, ακριβώς επειδή υπήρχε πρόβλημα τεχνικό, είχαμε γλιτώσει αρκετά χρήματα τότε που δεν είχαμε συνεδριάσει στο Στρασβούργο. Λοιπόν, η κυρία Γιάτεν Μάκη αναφέρθηκε στο θέμα της αποτελεσματικότητας και εγώ όταν ψάχνω μερικές φορές ε, ένα έγγραφο στο γραφείο μου διαπιστώνω ότι το έχω στο άλλο γραφείο στην άλλη πόλη και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, με ενοχλεί. Ε, προφανώς και εγώ είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την σημερινή συζήτηση. Ε, ακόμα και αν ήμουν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι θα ήθελα να μην υπάρχει Στρασβούργο. Προφανώς ε, είμαι υπέρ του Westminster στο Λονδίνο, αλλά το να κάνει βόλτες στο Westminster, επειδή οι ψηφοφόροι μου ζουν προφανώς στο βόρειο τμήμα της χώρας, δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να δεκτώ. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ συνάδελφε. Εποφελούμε λοιπόν από την δυνατότητα η οποία μου δόθηκε, πολύ προσωρινά βέβαια, να προεδρεύσω τη συνεδριάσεως για να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου και να πω ότι πραγματικά μου έκανε τρομερή ε, θα έλεγα εντύπωση, αρνητική εντύπωση η η, αντιμετώπιση από πλευράς της κυρίας Γιατενμάκη του συμβάντος με τον αντιπρόεδρο Παπαστάμκο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δίνει ε, μάχη για τη ζωή και είναι εντελώς άσχετο με το θέμα που συζητάμε σήμερα. Ήταν απαράδεκτο που το θέσατε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα ο ε, Απερθών πρόεδρος ο κύριος Καζίνη και εγώ είμαστε οι μόνοι που είμαστε μέλη αυτού του κοινοβουλίου στη δεκαετία του 80. 84 με 89. Θέλω να σας πω λοιπόν, αφήνω το κόστος στην άκρη. Να σας θυμίσω μάλλον ότι η Γαλλία εθιμικά μόνο, το Στρασβούργο εθιμικά μόνο είχε την ολομέλεια του Κοινοβουλίου ότι όταν αποφασίστηκε να γίνει κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες η Γαλλία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τότε ορίστηκε ως έδρα το Στρασβούργο ενώ ήδη οι συνθήκες από την αρχή όριζαν ως έδρα της Γραμματείας το Λουξεμβούργο. Από τη στιγμή που ορίστηκε ως έδρα το Στρασβούργο η Γαλλία εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια διευκόλυνσης των βουλευτών στο έργο τους. Κυρία Λεγκρίπ, το 1999 ήμουν πάλι μέλος αυτού του κοινοβουλίου και θυμάμαι τον πρόεδρο Σιράκ ο οποίος ήρθε στην Ολομέλεια και ομολόγησε ενώπιον όλων ότι η Γαλλία είχε εγκαταλείψει το Στρασβούργο κύριος Ντάφ ήταν εκεί ότι δεν κάνει αυτό που γινόταν στη δεκαετία του 80 και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Να σας τα πω πολύ απλά δηλαδή. Πράγματι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράζει την πολυμορφία των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν αυτή τη στιγμή υπήρχαν οι διευκολύνσεις που υπήρχαν στη δεκαετία του 80, δηλαδή αεροπορικές πτήσεις, δηλαδή η δυνατότητα μέσω της, ε, ε, της Δημαρχίας του Στρασβούργου να εξυπηρετούνται οι βουλευτές, οι επισκέπτες, οι πολιτικές ομάδες κτλ να μπορούμε να ταξιδεύουμε παραδείγματο χάρη μέσω Ελβετίας, κάτι που τώρα δεν μας το επιτρέπει το Κοινοβούλιο, και να υπάρχουν πτήσεις. Κύριε Καζίνη, για σας μιλούσα, έλεγα ότι εγώ και εσείς είμαστε στη δεκαετία του 80 εδώ και ξέρουμε τι γινόταν. Εάν λοιπόν δεν αποφασίσει η πόλη του Στρασβούργου να συμπεριφέρεται ως ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, θα έχουμε συνεχώς αυτά τα προβλήματα. Και εμείς που θέλουμε αυτή την πολυμορφία και δεν θέλουμε να είναι η Γαλλία εκτός και θέλουμε να διατηρηθεί το Στρασβούργο, είμαστε πάρα πολύ ενοχλημένοι από αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή από την απίστευτη ταλαιπωρία για να έρθουμε μέσω Φραγκφούρτης, να μην μπορούμε να φύγουμε σε άλλη μέρα ενδιαμέσως, να μην μπορούμε να έρθουμε τρίτη πρωί αν κάτι συμβαίνει στη χώρα μας και θέλουμε να μείνουμε εκεί. Ή λοιπόν θα αποφασίσει το Στρασβούργο την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα ή εγώ δεν το βλέπω καλό το μέλλον. Δηλαδή ακόμη και εμείς οι οποίοι επιμονή μου βάσεως ψηφίζαμε πάντοτε για τη διατήρηση του Στρασβούργου έχουμε αρχίσει κυρία Λεγκρίπ να έχουμε πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Λοιπόν, επανέρχομαι, δεν ήσασταν εδώ και θυμίζω τι είχε πει ο πρόεδρος Σιράκ και τι είχε υποσχεθεί. Πρέπει το γαλλικό κράτος να κάνει κάτι και όχι να έχει ένα περιφερειακό αεροδρόμιο που ανήκει στο Chamber of Commerce και λειτουργεί δηλαδή σαν να είναι μία μικρή επαρχιακή πόλη της πατρίδας μου που δεν έχει καμία σχέση με περιφερειακή χώρα. Επομένως για μένα δεν είναι θέμα οικονομικό. Της δημοκρατίας τα έξοδα πρέπει να τα πληρώσουμε. Είναι θέμα αποκλειστικά ρύθμισης ορισμένων πραγμάτων ώστε να μην είναι τόσο επιβαρυντικό το Στρασβούργο για τους βουλευτές και τους συνεργάτες τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μορέιρα. Το θέμα της έδρας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα το οποίο συνταγματικά ορίζεται από ένα συγκεκριμένο διακρατικό πρωτόκολλο. Προφανώς το Κοινοβούλιο έχει την δυνατότητα να προτείνει τροπολογήσεις στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Εγώ είμαι υπέρ ε, της ενιαίας έδρας εργασίας του Κοινοβουλίου και το δηλώνω αυτό σε αιτήσια βάση όταν συζητάμε το θέμα του προϋπολογισμού. Δεν έχει νόημα να έχουμε την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και το Κοινοβούλιο αλλού. Η άποψή μου λοιπόν είναι σαφής. Ε, δεν θέλω να αντιπαρατεθώ, αλλά ε, όπως είπα διαφωνώ με αυτούς που πιστεύουν ότι μπορεί να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, ε, το έχουμε ξανασυζητήσει σε διάφορες συνεδριάσεις. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τη συνθήκη της Λισαβάνας. Ε, έχουμε υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη, δεν έχει νόημα. Έχουμε 756 και 751 βουλευτές. Ε, έχουμε θέμα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Κοινοβουλίου καταρχήν. Ε, νομίζω ότι το να έχουμε δύο έδρες και να είμαστε μακριά από την διακυβέρνηση της Ένωσης δεν βοηθάει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εργασίας του Κοινοβούλου. Δεύτερον, ότι η θυσία που κάνουν οι ευρωβουλευτές όσον αφορά την μετα... τα ταξίδια, κατά... τα καταλήμματα κτλ. Δεν νομίζω πως αξίζει τον κόπο για να κάνουμε τόσο μεγάλες θυσίες. Τρίτον, είναι η δαπάνη, η σπατάλη ε, πόρων. Αλλά δεν είναι το τελευταίο επιχείρημα, είναι το τρίτο. Ε, δεν είναι μάλλον το πρώτο επιχείρημα, είναι το τρίτο. Γι' αυτό το λόγο ε, υπάρχει αυτή, η διαμάχη. Ε, υπάρχουν θέσεις των ευρωπαϊκών ε, κομμάτων, αλλά των ομάδων, αλλά και έχουμε και προσωπικές θέσεις ο καθένας. Εγώ ε, πιστεύω πως ε, ε, μπορούμε να πούμε ότι τέλος ε, από τη μια μέρα στην άλλη το Στρασβούργο πρέπει να υπάρξει κάποια αποζημίωση για τα κτίρια, για τα πλονεκτήματα των οποίων χαίρεται το Στρασβούργο με κάποιο τρόπο θα πρέπει να συνεχιστεί εκεί να δοθεί μια αποζημίωση. Το κάνω και εγώ μια πρόταση να, χωρίς να θέλω να είμαι προκλητικός, να μεταφερθούν στο Στρασβούργο η έδρα της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Δεν θα χάσουν τίποτα αν μεταφερθούν εκεί. Το να είναι μακριά από την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αλλάξει τίποτα στη λειτουργία τους και νομίζω πως είναι ένας δίκαιος τρόπος για να αποζημιωθεί η Γαλλία και το Στρασβούργο εάν αποσυρθεί από εκεί το Ευρωκοινοβούλιο. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο μικρό χρονοδιάγραμμα, πιο σύντομο. Είναι σημαντικό το θέμα. αλλά δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόσο εκταμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορούμε να ψηφίσουμε τον Νοέμβριο μπορούμε ίσως να κάνουμε πιο σύντομα και να τελειώνουμε σε δυο τρει μήνες νωρίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Μορέιρα και τώρα ο συνάδελφος Σούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά ο συνάδελφος Κουτιέρη με οδήγησε στο να τον ζητήσω παρόλα αυτά. Συμφωνώ 100% όταν λέει ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ποσοτικά πόσο μας στοιχίζει η δημοκρατία. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, θα πρέπει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τι στοιχίζει αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, να δούμε αν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, πιο οικονομικά και όπως ξέρετε το 2014 είναι ένα έτος εκλογών και όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα το οποίο θα τους θέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και χρειαζόμαστε όντως μια βαθιά συζήτηση, μια σωστή επεξεργασία του θέματος, ένα χρονοδιάγραμμα που να μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί επαναλαμβάνω η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντολογική και οικονομική πτυχή και είναι κάτι που σαφώς θα πρέπει να το συζητήσουμε, το θέμα της κυριαρχίας, το αν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει μόνο του και το θέμα της μίας και μοναδικής έδρας μπορεί να απαντηθεί με έναν απλό πρακτικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ πιο περίπλοκο το θέμα από ότι αρχικά ε, θα θέλαμε να είναι. Ε, εμπλέκονται πολλοί φορείς, πολλοί και διαφορετικοί φορείς και είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια προσεκτική και εις συζήτηση. Τώρα το θέμα της νομοθετικής εξουσίας Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και αν θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ε, χώρο. Σήμερα, όπως είπατε, έχει αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Υπάρχει μια εξισορρόπηση και αναρωτιέμαι, θα μπορούσαμε να το δούμε και διαφορετικά το θέμα, το θέμα της διακυβερνητικής μεθόδου, το θέμα της μεθόδου αυτής και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος στο μέλλον, κατά την άποψή μου, θα τροποποιηθεί περαιτέρω. Ε, εδώ είναι το κεντρικό σημείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τι προοπτικές θα έχουμε στο μέλλον και πώς μπορούν αυτές οι προοπτικές να γίνουν πιο ενισχυμένες, καλύτερες για μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει, συμφωνώ, οι προοπτικές όμως των περαιτέρω αλλαγών είναι αυτές που πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ε, ε, ε. Τρομακτικό είναι να είμαι τελευταίος ομιλητής. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φόξ που τόνισε ότι θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση ε, και τα γεωγραφικά θέματα έχουν σημασία. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε συνένεση είναι να έχουμε μία μόνο έδρα αντί να έχουμε 27. Τόνισε τρεις λόγους για τους οποίους θα μπορούσαμε να το στηρίξουμε αυτό και θα στοιχημάτιζα ότι αν αρχίσουμε να ψηφίζουμε στην Ολομέλεια για το Στρασβούργο ή για τις Βρυξέλλες θα ήταν 600 υπέρ των Βρυξελών και οι υπόλοιποι υπέρ του Στρασβούργου και εγώ μέσα σε αυτούς τους 600. Καταλαβαίνω γιατί είμαστε έτσι ταπεινοί. Ε, ξέρουμε τα όρια μας. Όταν όμως πρόκειται για το Συμβούλιο και την ομοφωνία που χρειάζεται εκεί, ο μόνος τρόπος είναι να πάμε στο Στρασβούργο και να σταματήσουμε τις δραστηριότητε στις Βρυξέλλες. Γιατί σε εκείνη την περίπτωση δεν χρειάζεται καν αλλαγή συνθήκης. Και τώρα η συνθήκη η ίδια πρέπει να αλλάξει ε, από πολλές απόψεις. και όχι μόνο στο πλαίσιο αυτού του όχι και τόσο θέμα θέματος της μιας έδρας, ίσως να προκύψει και το θέμα λοιπόν, της αλλαγής της συνθήκης. Γιατί αν μείνουμε σε ταπεινούς ε, και μετριοπαθείς στόχους, στο χαμηλότερο δηλαδή κοινό παρανομαστή, δεν θα πετύχουμε τον ρόλο που πρέπει για το Ευρωκοινοβούλιο. Και τώρα όσον αφορά τα κόστη. Εκτιμάται ότι είναι 200 εκατομμύρια ετησίως για πηγαίνω ερχόμαστε με όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ μας. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, το κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ορμήξει κάθε φορά. Και ο και στη χώρα μου το κοινοβούλιο δεν μετακινείται. Όποιο θέλει να δει κάποιον από το κοινοβούλιο έρχεται να τον δει εκεί. Άρα λοιπόν εμεί πάμε στο Στρασβούργο θα πρέπει να έρχεται η Κομισιόν να έρχεται στο Στρασβούργο. Η εικόνα του Κοινοβουλίου λοιπόν υποφέρει λόγω όλων αυτών. Και τέλος, ας φανταστούμε ότι θα περάσει η στήριξη για τη μία έδρα και κατά συνέπεια θα έχουμε αυτό το θέμα. Πού θα είναι αυτή η έδρα? Να το συναποφασίσουμε. Μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα. <laughs> και να σας ρωτήσω, όχι μόνο οικονομικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά, αλλά και αισθητικά. Το Στρασβούργο είναι πιο όμορφο από το Στρασβούργο. Που έχει, από το, Στρασβούργο είναι πιο όμορφο από τις Βρυξέλλες. Που οι Βρυξέλλες έχουν ωραία μέρη, ωραία σημεία, αλλά άλλα σημεία αλλά είναι σαν να βρίσκεσαι και να περπατάς μέσα σε ένα εφιάλτη, ακόμα και στις πόλεις του Έρικ Χόνιχερ. Και τώρα θα απαντήσουν οι συγητές, οι δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν αντίστροφα. Ε, ο συνάδελφος Έφνερ είχε πει ότι εκείνο θα έκανε ε, το, την τελευταία ομιλία. Ναι, ναι. Είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες για αυτήν την πρώτη ανταλλαγή ε, με τους συναδέλφους. Είδατε κι εσείς, διαπιστώσατε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις Όλες όμως θα εκπροσωπηθούν. Είναι όμως ένα καλό σημείο κίνησης αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα. Ακούστηκαν ουσιαστικά σημεία, σημαντικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Εμείς εκφράσαμε την άποψή μας λέγοντας ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά όχι άσκοπος χρόνος. Θα επεξεργαστούμε λοιπόν τις πρώτες προτάσεις και θέλουμε στις αντιπροσωπείες, στα πολιτικά κόμματα, στις πολιτικές ομάδες να συζητηθεί το θέμα, να κινητοποιηθούμε όλοι. Οι κυβερνήσεις να εμπλακούν έτσι ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε το θέμα αυτό να καταλήξει σε αδιέξοδο. Και να βρεθεί τρόπος, αυτή είναι η επιθυμία μας, με επικοδομητικό τρόπο να προχωρήσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βιαστούμε υπερβολικά να αφαιθεί ο απαραίτητος χρόνος για να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Θα υποβάλουμε λοιπόν το πρώτο σχέδιο με αρκετό υλικό έτσι ώστε να μπορέσετε να βασιστείτε σε αυτός. Θα οργανωθεί και η πρώτη ακρόαση. Να δοθούν κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που θα έχουμε θέσει. Η πρώτη έκθεση θα είναι έτοιμη μετά την ακρόαση του Μαΐου τον Ιούνιο. Για την επόμενη δηλαδή συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα ακολουθήσουν οι τροπολογίες, θα συζητηθούν τον Ιούλιο στην Επιτροπή οι τροπολογίες και κατόπιν βάσει όλων αυτών θα υποβληθούν συμβιβαστικές τροπολογίες το Σεπτέμβριο στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις μεταξύ των σκιωδών και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην προβλεπόμενη ημερομηνία εδώ στην Επιτροπή. Αν ε, διατηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες διαπραγμάτευση συζήτησης και έκφρασης, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις όλων. Τώρα, τα άλλα σημεία που αναφέρατε. Για μας είναι γνωστή η κατάσταση από νομικής απόψεως, τουλάχιστον γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Τι λαμβάνουμε υπόψη μας και από εκεί ξεκινάμε. Το Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό το θέμα. Θα δούμε αργότερα τα συναφή αν θέλετε, ε, εμείς σαν κοινοβούλιο αναρωτιόμαστε γιατί πραγματικά κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά στους ψηφοφόρους μας το ερώτημα αυτό προκύπτει. Και εμείς λοιπόν σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Είτε ναι, μας ικανοποιεί αυτή η κατάσταση, είτε όχι, κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ λοιπόν σαν εισηγητής θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζουμε την νομική κατάσταση και την προϊστορία, την ιστορία και το γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Το ερώτημα είναι αν πρέπει αυτό να διατηρηθεί επάπειρον ή αν κάπου κάτι πρέπει να αλλάξει. Όλοι όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα τα στοιχεία αυτά που μας οδήγησαν σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Και ο Ρομπέρτο έθεσε πολύ σωστά ερωτήματα. Εμείς σαν κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφύγουμε ε, να εκφραστούμε για τα άλλα θεσμικά όργανα. Να κάνουμε προτάσεις, ναι, αλλά για το ίδιο το κοινοβούλιο. Σκοπός μας είναι, από τη δική μας άποψη τουλάχιστον, Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει αυτή η συντακτική συνέλευση μετά τις εκλογές. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα θέματα και είναι σημαντικό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε σε αυτήν την συνέλευση με συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα, αν προκύψει το θέμα της έδρας των άλλων θεσμικών ορμάνων από τις κυβερνήσεις ή από κάποιον άλλον, εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Ας το αφήσουμε σε άλλους αυτό. Και εμείς θα περιοριστούμε αποκλειστικά και μόνο στο θέμα που αφορά την έδρα του δικού μας θεσμικού οργάνου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή. Να δω τώρα τι άλλο άκουσα από εσάς, έχω σημειώσει. Κάτι που θεώρησα πολύ σημαντικό όταν άκουσα την κυρία Λεγκρίπ είναι ότι μιλήσατε για την ιστορική κατάσταση, την νομική και είπατε ότι το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουμε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ή ένα πολυκεντρικό μοντέλο, όπως είπατε. Μιλήσατε για την κινητικότητα, μιλήσατε για τα ταξίδια. Έτσι κι αλλιώς έχετε δίκιο, θα συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε. Είναι τμήμα της αποστολής μας. Το θέμα είναι η Επιτροπή, το Συμβούλιο έχουν την έδρα τους κάπου, πρέπει και εμείς να πλησιάσουμε. Είτε είναι πιο σημαντικό να υπάρχουν πολλά κέντρα όπως είπατε. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το απαντήσουμε, είναι μια ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση είναι αυτή που καλούμεθα να συζητήσουμε. Και δεν υπάρχει μία μόνο καλή απάντηση. Το θέμα του κόστους, βέβαια. Και όταν αναφέρομαι στο κόστος το οικονομικό, Αναφέρομαι και στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, στις επιπτώσεις για το περιβάλλον, στο κλίμα. Και συμφωνώ με τον Ρομπέρτο. Εδώ Βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Από την άλλη μεριά η δημοκρατία δεν μπορεί να μετριέται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Σούλτς όμως είπε ότι αυτά τα χρήματα που δαπανάμε δεν είναι δικά μας. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αν δηλαδή ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, ναι ή όχι, θεωρεί λογική αποδεκτή δαπάνη αυτήν τη συγκεκριμένη δαπάνη την οποία εμείς θεωρούμε απαραίτητη για τη δημοκρατία. Σημείωσα λοιπόν όλα όσα είπατε, μην ανησυχείτε. Θα επανέλθω σε όλα αυτά που είπατε, κύριε Κάραντ, και τα δικά σας, τα σχόλια. Μιλήσατε για το αισθητικό κομμάτι του Στρασβούργου, την ομορφιά αυτής της πόλης. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας. Για μένα, όταν ταξιδεύω, ακόμα και όταν πήγαινα στις ε, πρώην σοσιαλιστικές χώρες, και είχα φίλους που σπούδαζαν εκεί στις χώρες του ταρκτού ε, σοσιαλισμού. Και πολλές φορές αυτό που πάντα με εντυπωσίαζε είναι η έλλειψη αισθητικής. Και έλεγα αυτό το σύστημα σίγουρα απέτυχε στο αισθητικό του κομμάτι. Για μένα λοιπόν το θέμα της αισθητικής είναι σημαντικό και για τη δημοκρατία και για ένα κοινοβούλιο. Θα το λάβω λοιπόν υπόψη μου και αυτό. Θα ήθελα λοιπόν και εξ ονόματος ε, του συναδέλφου Φόξ να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους παρόντες και μη να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια κοινή θέση. Να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν, γιατί πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα είναι σαφές ότι όταν ελήφθη η απόφαση να ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πήρε την απόφαση από μόνο του. Η απόφαση λήφθη στο Συμβούλιο. Και εμείς καλούμεθα σήμερα να απαντήσουμε αν όλα πρέπει να παραμείνουν όπως είχαν αποφασιστεί τότε ή αν κάτι πρέπει να αλλάξει. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη σήμερα, απόφαση θα πρέπει λοιπόν ίσως να μπορέσουμε να ξαναδούμε και το θέμα της έδρα μας. Και το ίδιο ισχύει και για την ημερήσια διάταξη και για το χρονοδιάγραμμα και για το πώς και πού θα συνεδριάζουμε. Ωραία, ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν. Ο κύριος ε, Φόξ δεν θέλει να παρέμβει. δύο λόγια. Λοιπόν, να μετρήσουμε την απόδοση, να μετρήσουμε το κόστος και να μετρήσουμε και την ε, ομορφιά υπάρχει κόστος, κόστος ε, θα πρέπει να θυμίσουμε όλες τα μνημεία, όλα τα βγούμε με μια ισορροπία, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα σε όλε αυτέ τι αξίε. Σημείο 13, ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματο Στοκχόλμη, για το οποίο είμαι εγώ εισηγητή. Μπορούμε να το ήσυχα-ήσυχα να το αναβάλουμε ε, γιατί είναι μια ανέκθεση που έχουμε το, με βάση το άρθρο 51 μαζί με την Επιτροπή Λίμπε και τη Γιούρη. Και το μόνο θέμα είναι ότι εγώ υποστηρίζω τη θέση ότι πριν να δώσουμε ένα έγγραφο θα πρέπει να γνωρίζουμε από την Κομισιόν ποια είναι η δική της θέση για την ενημέρωση, μάλλον την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ποιες είναι οι προοπτικές ε, που, για να τα αφήσουμε για την επόμενη θητεία. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να προηγηθεί μια ερώτηση προς την Κομισιόν από όλους τους συζητητές μαζί λοιπόν και μετά να παρουσιάσουμε το έγγραφο. Και έτσι μπορούμε να κλείσουμε τις εργασίες μας. Να θυμίσω ότι η τακτική μας συνεδρίαση προβλέπεται για τις 22 Απριλίου στις, ε, στις 3 και έπειτα την επόμενη μέρα 23 Απριλίου στις 9. Αλλά πριν στις 15 θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση για να ψηφίσουμε για την ε, έκθεση για τη για τα κόμματα.